Ευχθεί αύριο στις 12.30. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για προφορική ερώτηση Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ε, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Αρλέν Μακάρθη, που είναι συντάκτης, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την προφορική ερώτηση. Ακριβώς την καταθέσαμε για να γίνει ε, πρόοδος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαμεσολάβηση ε, με τον τρόπο που την ε, γνωρίζουμε, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, ε, μπορεί να εξοικονομήσει και χρόνο και χρήμα, γιατί κοστίζει η δικαστική οδός. Το 70% στην Ευρώπη επιτυγχάνει αυτή και 80% εάν την επιλέξουν εγκαίρως η διάδικη. Σήμερα όμως μόλις το 1% το επιλέγει. Η εμπειρία από τη δική μου χώρα είναι ότι ε, είναι πολύ δαπανηρή, 51.000 ευρώ η δίκη κατά μέσο όρο, είναι διαμεσολάβηση περίπου 87 ημέρες το 1 τρίτο και ένα κλάσμα του κόστους 9.000 ευρώ. Το 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας λέγουν ότι δεν δίνουν ε, συνέχεια ε, σε μια αγωγή σε ένα άλλο κράτος μέλος αν είναι το κόστος χαμηλότερο από 50.000 ευρώ γιατί τελικά ε, θα τους ε, φύγουν όλα τα λεφτά στα δικαστήρια και δεν θα πάρουν πίσω τις ε, αποζημιώσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πώς έχει η κατάσταση κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι. Η κατάσταση είναι και απογοητευτική και μας προβληματίζει. Βλέπουμε ότι ακόμα και η μικρή επιτυχία ε, ε, στη διαμεσολάβηση μπορεί να σημαίνει εξοικονόμηση και χρόνου και χρήματος. Αλλά ο κόσμος δεν προσφεύγει σε αυτή τη δυνατότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ε, δεν είναι πρόθεση των τριών θεσμικών οργάνων. Στο άρθρο 1 λέμε ότι ο βασικός στόχος οδηγίας είναι να επιτυχάνεται και να διευκολύνεται η διαμεσολάβηση, η εξοδικαστική και εναλλακτική επίλυση διαφορών ε, με φιλικό διακανονισμό και να δημιουργηθεί μια ισόρροπη σχέση μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών. Δηλαδή τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, δρά ε, και μάλιστα με ταχύτητα για να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ επίγον αυτό σε περίοδους ύφεση, σε περίοδους λιτότητας, σε περίοδους που τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να προωθούν τις οικονομίες χρόνου και οικονομίες χρημάτων. Έρχομαι στην ερώτηση λοιπόν. Κύριε Επίτροπε, πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα για να γίνει πρόοδος διότι δεν ε, πληρούνται ταχαίως οι ε, στόχοι της οδηγίας και συγκεκριμένα πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διασφαλίσει ότι πράγματι τη ισόρροπη σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και διαδικαστικών, δικαστικών, συγγνώμη, Θεωρεί ότι αυτή η επέτηση ε, να έχει την υποχρέωση των κρατών μελών να θέσουν και να επιτύχουν ένα ελάχιστο ποσοστό υποθέσεων στις οποίες χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα, τουλάχιστον όσον αφορά τις διασυνοριακές διαφορές. Και αν αυτό συμβαίνει, τι είδου μέτρα σκοπεύει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που αυτό το ελάχιστο ποσοστό δεν έχει τεθεί ή δεν έχει επιτευχθεί. Χαιρόμαστε για την ευκαιρία που έχουμε ε, να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σημαντικό θέμα. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Κομισιόν η Αντιπρόεδρος κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με την συντάκτρια της προφορικής ερώτησης γιατί η διαμεσολόβηση όντως είναι ταχύτερη και γενικώ είναι και φθηνότερο μέσω διακανονισμού των διαφορών από ότι μια δίκη στο δικαστήριο και επίσης δημιουργεί ε, μία ε, συμπεριφορά αποφυγής ε, της δίκης. Γιατί στην στη δίκη, οι διάδικη είτε μπορεί να είναι νικητές είτε ιτημένοι. Δημιουργείται αντιπαράθεση. Ενώ στη διαμεσολάβηση υπάρχει συνεργασία. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια πεδία διαμεσολάβησης που είναι πολύ πιο θετική. Τώρα πώς θα το καταφέρουμε. Η διαμεσολάβηση και η σχετική οδηγία υιοθετήθηκε το Μάιο του 2008 και θα έπρεπε να μεταφερθεί την 21η Μαΐου του 2011. Βέβαια όλα τα όλα τα κράτη-μέλη είναι θετικό ότι έχουν ήδη κοινοποιήσει τα μέτσα για την εσωμάτωση της οδηγίας. Μετά από ένα χρόνο μόνο εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη-μέλη, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο και δεν έχουμε συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα ε, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα κατά πόσο τηρήθηκε ή όχι οδηγία. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Και για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες θα καταθέσουμε και ανακοίνωση για τη διαμεσολάβηση τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2013, προκειμένου να προωθήσουμε τη χρήση της διαμεσολάβησης. Και στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνουμε και εκτεταμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία και την χρήση της οδηγίας από τα κράτη-μέλη. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στη σημασία που έχει η προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου επίλυσης των διαφορών. Γιατί ε, αν, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφέρουσα νομοθεσία, αλλά κανένα δεν τη γνωρίζει, γιατί μερικέ φορέ δεν τη χρησιμοποιούν ούτε οι δικαστέ ούτε οι δικηγόροι, τότε είναι σαν να μην υπάρχει. Πρέπει λοιπόν ε, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη σχέση μεταξύ της ε, διαμεσολάβηση και της ε, δίκη, της διαδικασία σε δικαστήριο. Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί πολύ περισσότερο ε, και σε διασυνοριακέ διαφορές. Ω εκ τούτου ζητήσαμε στις εθνικές εκθέσεις που θα συγκεντρωθούν στα πλαίσια της μελέτης που εκπονούμε ε, καλό θα ήταν να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένες πληροφορίες για την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διαμεσολάβηση και των ε, δικαστικών διαδικασιών και των δικών στα κράτη-μέλη. Και με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα σκεφτούμε τι μέτρα θα προτείνουμε στο μέλλον για να ενισχύσουμε την προσφυγή στη διαμεσολάβηση και να επιτύχουμε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ διαμεσολάβηση και δικών. Τώρα, σύμφωνα με την οδηγία, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο, δεν κομίζω βλάπιες Αθήνας, θα υποβληθεί και έκθεση το 2016 και με βάση την έκθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο η οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί, να αναθεωρηθεί, να εμπλουτιστεί με νέες προτάσεις. Πάντως, στο μεταξύ, πιστεύω ότι δεν θα περιμένουμε την έκθεση του 2016. Έχουν στο μεταξύ υποβληθεί και άλλες προτάσεις και θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρόλα αυτά. Γιατί η, μεθολα... η διαμεσολάβηση θα πρέπει να θεωρηθεί και στα πλαίσια του προγράμματός μας δικαιοσύνη για ανάπτυξη. Ξέρετε ότι έχουμε συνδυάσει πολλά μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως τις διασυνοριακές ε, εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χάρη σε κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαιωτικό σύστημα και η διαμεσολάβηση είναι μία από αυτές τις μεθόδους και μάλιστα στην ετήσια έκθεση ε, για την ανάπτυξη του 2013 που η αρχή της προτεραιότητες για τη μεταρρύθμιση περιλάβαμε ως προτεραιότητα και τη διαμεσολάβηση. Και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα κατάλογο επιδόσεων σε θέματα δικαιοσύνης και θα αναλύσει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες του δικαιωτικού συστημάτων των κρατών μελών. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο από τα κράτη-μέλη για να ενισχυθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία του, προγρά... του συστήματος των αστικών δικαστηρίων γιατί η ποιότητα, η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη ή μπορεί να καταπνίξει την ανάπτυξη. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη στην ετήσια επισκόψη της ανάπτυξης και ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθεί η χρησιμοποίηση τη διαμεσολάβηση στα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα να επιτευχθεί χάρη σε, κατάρτιση, σε κατάλληλη κατάρτιση, ενημέρωση και συνειδητοποίηση των πολιτών ότι η διαμεσολάβηση είναι ενδιαφέρον τρόπος επίλυση των διαφορών. Ιστερούμε κάπως σε πρόοδο, γι' αυτό και πιέζουμε τα πράγματα για να σημειώσουμε ταχύτερα πρόοδο. Ευχαριστώ. Πολύ την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτη ομιλήτρια εξ ονόματος του ΕΛΚ είναι η συνάδελφος κυρία Ματσόνη. Για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ε, συμφωνώ τόσο με αυτά που είπε η κυρία Μακάρτη, όσο και με αυτά που είπε η Επίτροπος ε, κυρία Ρέντινγκ υπάρχουν αναμφίβολα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν εφόσον έχουμε μια αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαμεσολάβησης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε αρνητικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να συνεχίσουμε τους ελέγχους γιατί μόνο εδώ και ένα χρόνο ε, έχει εκπνεύσει ο χρόνος ε, κατάθεσης προτάσεων. Αν κρίνουμε από την Ιταλική εμπειρία, ε, νομίζω ότι πρέπει να παρατηρήσουμε περαιτέρω την όλη υπόθεση, γιατί εμείς ε, είχαμε, διαπιστώσαμε κάποια εξοικονόμηση, περίπου 480 εκατομμύρια ξεκονομήσαμε σε ένα χρόνο εφαρμόζοντας ε, τις διαδικασίες αυτές σε 49% των περιπτώσεων. Άρα δηλαδή ιδιαίτερα θετικό. Ας δούμε λιγάκι τα αρνητικά στοιχεία. Αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι ότι έχει ξανανοίξει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο στη χώρα μας μία απόφαση που αναφέρει ότι υπάρχει αντισυνταγματικότητα ως προς την δεσμευτική εφαρμογή της ε, διαμεσολάβησης. Το 361 του 2011, αυτή, αυτός είναι ο αριθμός της απόφασης, αυτό το είπε σήμερα και η Επίτροπος, είπε ότι θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση του εργαλείου του μέσου της ε, διαμεσολάβησης Βέβαια αυτό είναι διαφορετικό από τη δεσμευτικότητα. Δηλαδή η Επίτροπος λέει κυρίως ότι θα πρέπει η διαμεσολάβηση να είναι εθελοντική και θέλω να γνωρίζω κατά πόσο αυτή είναι πραγματικά η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μήπως η Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη, μήπως πιστεύει δηλαδή ότι η δεσμευτικότητα έχει άμεση σχέση με τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, κάτι το οποίο πάλι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο δικαστής. Κυρία Ματσόνη, Εξ ονόματος της ομάδος S&D το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Σίλβια Αντριάνα Τικάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και Πρόεδρε. Ε, όντως είναι γρήγορη λύση, διαμεσολάβηση και φθηνή για ζητήματα εμπορικά και αστικά ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν ε, τη ε, διάθεση ενημέρωσης και στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό, την ύπαρξη διαμεσολαβητών και ποιοι προτείνουν τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης είναι σημαντική η εμπιστευτικότητα και το απόρριτο. Θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης δυνατότητα εξασφάλισης εχεμήθειας σε αυτή την προσπάθεια. Κυρία Επίτροπε, ε, προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ενδιάμεση έκθεση πριν το 2016 για την εφαρμογή της Οδηγίας 52 του 2008. Θα θεσπίσετε κοινού ε, κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με προγράμματα κατάρτισης ενιαία παντού για να έχει κανείς πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή, να είναι καλύτερης ποιότητας η διαμεσολάβηση ε, και γενικότερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή είναι ο συνάδελφος κ. Κρίστιαν Σίλβιο Μπουσόη, εξ ονόματος ομάδος Άλτε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διαμεσολάβηση σε θέματα αστικά και εμπορικά και σε γενικότερα εξοδικαστική επίλυση των διαφορών είναι πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική και για τα ενεχόμενα μέρη αλλά και το δικαστικό σύστημα, ιδιαίτερα σε πολλά κράτη-μέλη όπου η δικαιοσύνη ε, είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιβαρημένη ε, από τις υπερβολικές δίκες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και θα πρέπει να τίθεται σε ισχύ όσο γίνεται καλύτερα. Η οδηγία για τη δημοσιολάβηση δεν έχει ακόμα επιτύχει τους στόχους ε, σε ό,τι αφορά το κλάσμα των ε, περιπτώσεων που καταφεύγουν στη διαμεσολάβηση και όχι στη δικαιοσύνη. Γιατί γίνεται αυτό, διότι ο κόσμος δεν το ξέρει ότι υπάρχει. Η οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση ενημέρωση του Εβραίου κοινού για τη δυνατότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ε, οι πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της διαμεσολάβησης, γι' αυτό και δεν τη χρησιμοποιούν. Δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες και επίση δεν ξέρουν σε ποιον αποταθούν για να κινήσουν τη διαδικασία αυτή. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο, τα εμπορικά ζητήματα, η νέα οδηγία ε, για την εναλλακτική εξοδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών θα φέρει μεγάλη πρόοδο, γιατί οι έμποροι θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πελάτες για τους ανακτικούς μηχανισμούς και τη διαμεσολάβηση. Ωστόσο, η οδηγία αυτή έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Άρα θεωρώ απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και τα κράτη-μέλη να κάνουν μεγαλύτερη διαφήμιση για αυτή τη δυνατότητα, ιδιαίτερα τη διασυνοριακή και το οικογενειακό δίκαιο. Εδώ εμείς δεν θέλουμε να χτίσουμε ένα σύστημα παράλληλο με το δικαστικό. Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να παραμένει μια δυνατότητα και να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στη δικαστική επίλυση και την εξοδικαστική. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε στόχους ε, ποσοτικούς και ποσοστιαίου για το πόσες ε, υποθέσεις θα πρέπει να καταλήγουν σε διαμεσολάβηση. Θα πρέπει πάντως να προωθήσουμε τη κουλτούρα της ενελικτικής επίλυσης διαφορών και της εξοδικαστικής. Είναι και πιο εύκολη και πιο γρήγορη και πιο φθηνή από τη δίκη και πραγματικό πλεονέκτημα για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουσόη. Ε, ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Σέρτζιο Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω και εγώ, όπως και η συνάδελφος Μακάρτη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να κάνει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να διδοθεί η πρακτική αυτή της διαμεσολάβησης. Πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες για την Ένωση, πρέπει να προωθήσουμε εκπαιδευτικέ δράσεις, Ουσιαστικά πρέπει να δώσουμε ουσία σε μια επιλογή μακρόπνοη που να μπορεί να δώσει αποτελέσματα θετικότατα για όλα τα άτομα προς τα οποία απευθυνόμαστε. Μετά, όπως αναφέρθηκε, αυτή η διαμεσολάβηση γίνεται ακόμα πιο χρήσιμη σε μια περίοδο ύφεση όπου οι διαθέσιμοι πόροι ε, για τους πολίτες, οικογένειας έχουν περικοπεί κατά πολύ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κάτι που είπατε και είμαι ικανοποιημένο που το υπογραμμίσατε. Η διαμεσολάβηση αυτή είναι και μια πολιτισμική επιλογή. Είναι μια επιλογή που μπορεί να επιτρέψει στι περιπτώσει αυτέ τι εμπορικέ και πολιτικέ να ξεπεράσουν οι δικαστικέ διεργασίε και να σχηματιστεί μια συγκεκριμένη ιδέα για τη σχέση μεταξύ ατόμων που έχουν κάτι ε, για το οποίο θα, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν για να λυθεί διαφορά. Και αυτή η νοοτροπία μπορεί να επεκταθεί και στα πλαίσια των υποθέσεων εργασία η συντάκτη ε, της προφορικής ερώτησης, η κυρία Μακάρθι. Ήθελα σε αυτή τη διαδικασία απλώς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, την Επίτροπο διότι αφοσιώθηκε ε, στο θέμα, ε, ανέλησε την απάντηση, σε ακολουθεί ενεργό προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να ακούσω τι απαντήσει σε ευαισθητοποίηση για την κατάρτιση. Τα διάφορα κέντρα είναι κεντρικό σημείο για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Επίτροπο ε, να ενημερώνει την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τις συνεχιζόμενες εργασίες, να επανέλθει σε εμά, διότι θέλουμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό καθήκον, διότι στο τέλος, όπως πολύ συχνά βλέπουμε, ε, ο φόρτος εργασίας, οι υποθέσεις που κολλάνε στα δικαστήρια και τεράστια, τεράστιος κόστος δεν είναι υποφελή για τους πολίτες μας. Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ρέντι. Μάικ. Uh, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης είναι στέρηση δικαιοσύνης ε, και σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε πάρα πολύ μεγάλη στέρηση σε αυτό το τομέα, οπότε η διαμεσολάβηση είναι μία από τις δυνατότητες που παρέχεται, ούτως ώστε να απαλλαχθούμε από αυτό, αυτή την καθυστέρηση, κυρίως στις μικρότερες υποθέσεις, όπου δεν είναι απαραίτητο να περάσει κανείς από μακροσκέλη διαδικασία δικαστική. Αλλά βεβαίως η πρόσφαση στη δικαιοσύνη είναι θεμελιώδες δικαίωμα, Οπότε δεν πιστεύω ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να αντικαταστήσει απλώς ε, μια εκδίκαση υπόθεσης, είναι εναλλακτική. Αλλά για να γίνει η πραγματική εναλλακτική λύση πρέπει να γνωστοποιηθεί και όπως σωστά υπόθηκε Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο και γι' αυτό ε, για να μπορούμε πρέπει να δούμε πώς το άρθρο 9 θα εφαρμοστεί. Το άρθρο 9 των διατάξεων αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα ενθαρρύνουν με οποιοδήποτε τρόπο που θεωρείται ενδεδειγμένο την διαθεσιμότητα προς το ευρύ κοινό των πληροφοριών. Εκεί λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση. Και εμείς έχουμε κάτι στο κείμενο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρθρο 10, που λέει ότι θα διαθέτουμε στο κοινό πληροφορίες στα αρμόδια δικαστήρια, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές που κοινοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Άρα εδώ είναι συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να διατίθεται περισσότερες πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, κατάρτιση των διαμεσολαβητών και χωρίς την ε, κατάρτιση και των νομικών ε, να μην θεωρούν τη διαμεσολάβηση σαν κάτι που είναι αντίθετο προς τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Οπότε επανέρχομαι και στην αλλαγή της νοτροπίας ε, και αυτό είναι κάτι που δεν θα γίνει εν μία νυχτή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς να το επιδιώξουμε και γι' αυτό εγώ θα εκδώσω αυτή την ανακοίνωση το 2013 επί τη βάση των πληροφοριών που θα έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη και θα δημοσιεύσουμε αυτά τα στοιχεία και θα το ξανασυζητήσουμε και θα αναλύσουμε τα διάφορα προβλήματα στα διάφορα κράτη-μέλη και έτσι μπορεί να οδηγηθούμε σε πίεση ομοτήμων που αυτό τελικά θα οδηγήσει στο να αποδειχθεί ότι είναι μια ορθή εναλλακτική διαμεσολάβηση κυρίως για μικρές αξιώσεις, μικρές διεκδικήσεις, για διαφορές μεταξύ γειτόνων, για εργατικές διαφορές, για οικογενειακές διαφορές, ούτω ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορούν να λύσουν έτσι τα προβλήματά τους και βέβαια εκεί πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την άκρος επικοδομητική του θέση. Merci, ε, Madame la